Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 11η Ιουλίου, μέρα μνήμης των θυμάτων της φραγής της Σρεμπρένιτσα. Το λόγο έχει ο Υπουργός Βόντρα ε, για το Συμβούλιο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη Σρεμπρένιτσα. Όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν εφρικτή η σφαγή περισσότερων από 8.000 Βοσνίων. Σημάδεψε την Βοσνία Ζεγοβίνη, την πρώην Γεκοσλαβία αλλά και όλη την Ευρώπη. Αναμφίβολα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ε, αγριότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Κοιτώντα αναδρομικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ, πιο πολλά και πολύ νωρίτερα. Ήταν ε, ένα, μια αποτυχία της ε, διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για κάτι το οποίο μετανιώνουμε. Είναι ηθικό μας καθήκον και πολιτικό μας καθήκον να μην επαναληφθεί ποτέ η Σρεμπρένιτσα. Η δέκατη με επέτειος της ε, σφαγής της Ρεμπρένιτσας αποτελεί φόρο τιμής για όσους χάθηκαν και για τις οικογένειές τους. Τονίζεται ότι η συνεχή συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και Κοσλαβία αποτελεί βασικό, βασικός όρο για τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσαγωγή του Ράτκο Μλάντης θα ήταν ένα σωστός φόρος τιμής για τα θύματα της Ρεμπρένιτσα και θα συνέβαλε στην σταθεροποίηση και την επανασυμφιλίωση στην περιοχή. Γι' αυτό το Συμβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι δράστες των εγκλημάτων στις Ρεμπρένιτσα αλλά και στη Βοσνία Ερσεγοβίνη γενικότερα καθώς και στην υπόλοιπη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και ότι αυτοί οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και παραλλήλου σε όλη την ιστορία η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να επουλώσει τις ε, πληγές του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, παράγοντας ε, συνένωσης έφερε ευημερία και αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, βοηθώντας τα Βετικά Βαλκάνια να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία από τις βασικές προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας. Και η επανασυμφιλίωση είναι απαραίτητη για την ε, ένταξη και η επανασυμφιλίωση είναι δύσκολη αν δεν έχει αποδοθεί πλήρωση η δικαιοσύνη. Μετά από τόσα χρόνια έχει έρθει ο χρόνος να κλείσει η πληγή της Ρεμπρένιτσα. Ο Καραντίτσα απέδειξε ότι δεν υπάρχει τιμωρησία για τέτοια κτηνόδια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, ο Ράτκο Μλάντινς δεν έχει ακόμα προσαχθεί στην Χάγη. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κλείσουμε το παρελθόν και να αγκαλιάσουμε το μέλλον. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη για να το πετύχει αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου η Σρεμπρένιτσα από ένα τραγικό επεισόδιο της ιστορίας να μετατραπεί σε ένα μέρος όπου η ζωή παρέχει ευκαιρίες. Δεν κινούμαστε στο κενό, συνδυαζόμαστε με τοπικές δράσεις και τοπικές εντότητες. Έχουν γίνει και πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Η Σρεμπρένιτσα θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κόσμου στη Σρεμπρενίτσα. Οι αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας και της ε, Βοσνιακής ε, Αρχής παρέχουν χρηματοδότηση και επενδύσεις για την περιοχή. Τα κονδύλια αυτά αποσκοπούν στην ανα ανοικοδόμηση και την ε, ανάπτυξη υποδομών στην περιοχή, στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, στα σχετικά προγράμματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όλες αυτές οι προσπάθειες ε, ενισχύονται από συνεδρίαση δωρητών που διοργανώθηκε πριν από κάτι παραπάνω από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2007. Και ίσως είναι καλή ευκαιρία να απευθύνουμε μια έκκληση για εκ νέου χρηματοδότηση της περιοχής αυτής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Σερβρένιτσα να μην ξεχαστεί ποτέ και να συνεχίσουν οι κοινέ προσπάθειες. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα και οι τοπικές αρχές άλλωστε συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στην περιοχή της Ρεμπρένιτσα. Μόνο αυτή η προπτική της καλύτερης ζωής μπορεί να, αν θέλετε, απαλύνει τον πολιτική πίεση και τις πολιτικές εντάσεις, προκειμένου να επιτρέψει στα θύματα, στις οικογένεια των θυμάτων να προχωρήσουν. Αυτή θα ήταν, αυτός θα ήταν ο καλύτερος φόρος τιμής για τα θύματα της Ρεμπλένιτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επιτροπέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 1995 περίπου 8.000 ε, άνδρες ε, και παιδιά δολοφονήθηκαν στην Σαμπένιτσα. Όλοι κάλεσαν αυτήν την σφαγή ως γενοκτονία. Ε, ενώ συνεχίζεται η δίωξη των δραστών θα πρέπει να θυμηθούμε τα θύματα και να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στα της οικογένειάς τους. Γι' αυτό λοιπόν προστηρίζω την πρωτοβουλία να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως μέρα μνήμης των θυμάτων της φαγής Στρεμπρένιτσα. Η ιουλιου αποτελεί ένα σύμβολο της φρίκης και του πένθους. Η ανακήρυξη της επαιτίου είναι κάτι το απαραίτητο, διότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και χρειάζεται να τιμούμε την μνήμη των θανόντων. Τα αναγνώριση των όσων συνέβησαν τον Ιούλιο του 1995 είναι σημαντικό για τη συμφιλίωση στην Βοσνία Ριζεγοβίνη αλλά και στην ε, περιφερική διαδικασία. Το να ανακηρύξουμε την 10η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων της φαγής της Στεμπρέμιτσα θα πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς, περαιτέρω προς την συμφιλίωση επαναλαμβάνω, για την Βοσνία Ζεγοβίνη και για την περιοχή είναι, αποτελεί ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα όχι μόνο στη, για τη μνήμη των θανόντων αλλά και για ελπίδα για το μέλλον. Μια ελπίδα που θα βασίζεται στην ε, συμφιλίωση και να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές. Αλλά αναγνώριση δεν είναι ε, αρκετή. Η δικαιοσύνη είναι και αυτή απαραίτητη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι δράστες αυτών των φρικαλαιοτήτων να οδηγηθούν στα δικαστήρια, να δικαστούν και να πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Είναι λοιπόν απαράδεκτο ο στρατικός Ράτικο Μλάντιτς να είναι φυγόδικος. Η Κομισιόν ε, στηρίζει το έργο του Ίκτη του ποινικού δικαστηρίου για την Προϊκοσλαβία. Βοσνία Ερζεγοβίνη συνεργάζεται με το δικαστήριο και εμείς ως Κομισιόν χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να διασφαλίσουν πως όλα τα εγκλήματα θα διωχθούν. Κύριε Πρόεδρε, επιπλέον θα θέλαμε να Προσφέρουμε και μια δεύτερη μορφή δικαιοσύνη για τα θύματα, δηλαδή ένα καλύτερο μέλλον για τους επιζήσαντες, για τους αγαπημένου του. Αυτός είναι ένας σωστό τρόπος για να συμφιλειώσουμε την περιοχή. Θέλουμε να δούμε μια ευημερούσα Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο ενός σταθερού περιφερειακού πλαισίου όπου θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη Ξέρουμε ότι το ταξίδι αυτό θα είναι μακρύ, αλλά εάν η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διεύρυνσή της ε, μας διτάσχει κάτι, αυτό το κάτι είναι ότι το ταξίδι αξίζει για όλους τους εμπλεκόμενους. για να ολοκληρωθεί αυτός ο τρόμος θα πρέπει να εκπληρώσει τις ε, απαιτήσεις ε, και τα προαπαιτούμενα. Θέλουμε λοιπόν η Βοσνία Ζεγοβίνη να επιτύχει και να αποτελέσει το θρίαβο των επισάντων. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε ευχαριστώ. Για την ομάδα του ΕΛΚ το λόγο έχει η κυρία Πακ για δύο λεπτά. Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, Ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ ξανά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ποτέ ξανά γενοκτονίες. Μετά τις φρικαλαιότητες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί στην Ευρώπη ότι ξανά θα παρουσιάζονταν τέτοια φαινόμενα. Και παρόλα αυτά συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του 90, έξι χρόνια μετά την επιτώση του τείχους του Βερολίνου, στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Συνέβη ξανά. Τα ασφάλματα της διεθνούς κοινότητας μετά από πολλά χρόνια αγνόησης του προβλήματος της φιλικής διατηρήσης σχέσεων με τους εγκληματίες αυτούς ε, τους έκανε να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν ατιμόρυτοι να ξεφύγουν μετά από εθνοκαθάρσεις, μετά από γενεκτονίες, μετά από μαζικές δολοφονίες. Ως τώρα ο Μλάντης δεν έχει ε, συλληφθεί, ποιος τον κρύβει, ποιος τον καλύπτει. Πολλοί από τους εγκληματίες εξακολουθούν να είναι ασύλληπτοι, ακόμα και να μένουν στην ίδια τη Βοσνία Ζεγοβίνη και κοιτούν κατάματα, συναντούν καθημερινά τις οικογένειες των θυμάτων. Η επέτειος ε, θέλει να ανακοινήσει, να θέσει μία ένδειξη κατά της εγκατάληψης. Ίσως η ημέρα αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέρα που θα ξυπνήσει το υποσυνείδητο ακόμα και εκείνων που ακόμα δεν πιστεύουν ότι συνέβη αυτή η καταστροφή, που δεν πιστεύουν ακόμα και στις μαγνητοσκοπημένες φαγές. Χωρίς την αναγνώριση των άμεσα και έμεσα υπεύθυνων για την σφαγή αυτή δεν θα μπορέσει να υπάρξει ειρήνη. Αυτό τουλάχιστον και η καταδίκη των εγκληματιών είναι αυτό που οφείλουμε στα θύματα και στις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους των Σοσιαλιστών, ο κ. Χαουίτ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επέτειο των πολέμων του 20ου αιώνα χρησιμοποιούμε τις λέξεις κατά το ηλιοβασίλεμα και κατά την Ανατολή του ηλίου θα τους θυμόμαστε. Αυτές οι λέξεις πραγματικά με συγκινούν. Ακόμα και για τις γενιές εκείνες που μας ακολουθούν. Αυτή η μνήμη δεν αποτελεί μόνο ένα φόρο τιμής για αυτούς που έπεσαν. Μας υπενθυμίζει το όνειδος του πολέμου και αποτελεί και αν θέλετε μια δικλίδα για την ειρήνη για τα μελλοντικά χρόνια. Αυτό είναι η σημασία, αυτή είναι η σημασία της ε, επαιτίου και όπως είπε και η Επίτροπος, η αναγνώριση είναι πραγματικά κρίσιμη για την επανασυμφιλίωση για τις σημερινές γενιές. Όλοι ξέρουμε τις φαγές που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα το 1995. 8.000 μουσουλμάνοι, άντρες και αγόρια, σφαγιάστηκαν σε ένα δίθεν ασφαλές καταφύγιο στη Σρεμπρένιτσα. Παρόλο που αυτό συνέβη πριν από σχεδόν 14 χρόνια πλέον, είναι πρέπον και αρμόζουν να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα και να, να θυμηθούμε τα γεγονότα και το φλετικό μίσος που οδήγησαν στα γεγονότα αυτά. Τον προηγούμενο μήνα δημιουργήθηκε μια ομάδα χιλίων ατόμων στο Facebook που ανοιχτά βγήκε και ε, χειροκρότησε την ε, σφαγή της Ραμπρένιτσα. Η ομάδα αυτή επικρότησε τη σφαγή των ατόμων αυτών μόνο και μόνο επειδή ήταν ευώσνοι. Και η συνεχιζόμενη ελευθερία του Μλάντιτς αποδεικνύει ότι τον καλύπτουν αυτοί που προσπαθούν να καλύψουν τα γεγονότα του παρελθόντος. Χάρη στην ε, δημόσια κατακραυγή αποσύρθηκε αυτό το site στο facebook. Αλλά αυτό δεν είναι το γεγονός ότι έχει υπογραφεί από χιλιά άτομα. Η μνήμη των θυμάτων της Ρεμπρένιτσα αποστέλει ένα σαφές μήνυμα προς τα άτομα αυτά που ε, επικροτούν τις πράξεις του Μλάντης και όλων των υπόλοιπων εγκληματιών ότι δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ μαζί τους και ότι είναι απομονωμένοι Το βασικό πρόβλημα για πολλούς από τους ε, συγγενείς των θυμάτων είναι από ψυχολογικής άποψης ότι ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τους αγαπημένους τους. Πρόεδρε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας αυτής θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, από το Άλτερ, ο κύριος η Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε μια κοινή ιστορική μνήμη και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να οικοδομήσουμε κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Αυτό η Σρεμπρένιτσα αποδεικνύει ότι το έτος 1995 ε, επαναλήφθηκαν οι αγριότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Σρεμπρένιτσα αποτέλεσε σφαγή αθώων παιδιών, αθώων πολιτών. Και είναι φρικτή και η καταστροφή των μαζικών τάφων. Θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινή ιστορική μας μνήμη η Σρεμπρένιτσα. δεν επιτρέπεται να αποδεχτούμε αυτή τη στάση κατά κάποιων εθνοτήτων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη συλλογική αυτή ευθύνη και οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα της Ρεπρενίτσα θα πρέπει να προσαχθούν στη Χάγη, θα πρέπει να φυλακιστούν, θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τους πολίτες της Βοσνίας Ρεσεγοβίνης. και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα άτομα αυτά που ζουν με τη μνήμη των εγκλημάτων αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο που ομόφωνα συμφώνησαν για την ε, συμμετοχή και την πρόσκληση Βοσνίων στο Ευρωκοινοβούλιο κάθε χρόνια όπου από κοινού μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας. Ο κύριος ε, Χωρατσέκ, εκ μέρους των Πρασίνων. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα χρησιμοποιεί ξεκάθαρα λόγια. Οι μηχανισμοί στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να αποτρέψουν τα φρικτά γεγονότα στη Σεμπρένιτσα. Ως σήμερα η έλλειψη μιας κοινή φωνής αποτελεί ε, μια, ένα έλλειμμα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Μιλώντας για την σύραξη στη Γάζα, αυτό αποδείχθηκε εκ νέου. Η σφαγή στη Σρεμπρενίτσα δεν θα πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Γι' αυτό καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία για την καθιέρωση της 11ης Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενεκτονίας της Τρεμπλένιτσα. Εκ παραλλήλου θα πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση των δύο πλευρών. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επεξεργασίας των όσων συνέβησαν. Είναι απόλυτα απαράδεκτο η υπεύθυνοι των εγκλημάτων αυτών να εξακολουθούν να παραμένουν ασύλληπτοι. Νομίζω ότι όχι μόνο ο Μλάντιτς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσαχθούν στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξενόμαρος της ΓΚΟΕ, ο κύριος Μέγερ, το λόγο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, το όνομα της Ρεμπλιανίτσα έγινε παγκόσμια γνωστό λόγω των μαζικών ε, δολοφονιών 8.000 μουσουλμάνων το 1995 και δικαίως οι γυναίκες που επέζησαν μας καλούν να προσέξουμε το θέμα αυτό. Μετά την επίσκεψή μου στη Σραμπρένιτσα το Μάρτιο του 2007 ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει σε βιώσιμες λύσεις και θέσεις εργασίας στην πρόθεση του τουρισμού προκειμένου η Σρεμπρένιτσα να, έχει, να προσφέρει παραπάνω πράγματα από την ιστορία της. Η Σρεμπρένιτσα αποτελεί επίσης ένα σύμβολο της αποτυχίας των αισιόδοξων προοπτικών, των ανθρωπαστικών ε, εγχειρημάτων. Θα πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι η παρουσία ε, αλλοδαπών στρατευμάτων δημιούργησε μόνο λανθασμένες ε, προσδοκίες. Χωρίς τις Ολλανδικές δυνάμεις στη Σραμπρένιτσα δεν θα είχε προκύψει πόλεμος και δεν θα υπήρχαν τα συνεπακόλουθα. Δεν είναι μόνο απαραίτητο να... Θα πρέπει να σκεφτούμε διακόπτει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέλτερ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που σας... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένας ε, Βόσνιος με αγκάλιασε και έκλεψε και είπε «Σκοτώστε με μένα, γιατί σκοτώσατε και το παιδί μου. Δεν θέλω τίποτε άλλο, σκοτώστε με και εμένα». Αυτά αναφέρει μία Βόσνια γυναίκα, η οποία βρέθηκε στις Ρεμπλένιτσα το 1995 και έχασε και το γιο της, το 12χρονο γιο της και τον άντρα της. και ακούμε πολλά σχετικά στις κατοχώρες. Ναι, μεν προβάλλεται η ευρωπαϊκή προοπτική στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, αλλά θα πρέπει να τηρούμε και αυτή τη μνήμη για όλους όσους επέζησαν τις γενοκτονίες αυτής. Ρεμπρένιτσα 95. Παρακολούθησα την κατάσταση από κοντά και αισθάνθηκα πραγματικά ντροπιασμένο για την ε, αντίληψη του Safe Haven. Ως Ολλανδός πολίτης Γνωρίζουμε πάρα πολλούς ποιητές που έχουν γράψει σχετικά ποίηματα για τις ε, γενοκτονίες της Στοιανοφ. Ευχαριστώ κύριο Στογιάννοφ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να θυμηθούμε ένα φοβερό έγκλημα, μια γενοκτονία, μια τραγωδία στην πρόσφατη μας ιστορία. Διαβάζοντας όμως το σχέδιο ψηφίσματος, αυτό που προτείνεται, βλέπω ότι δείχνει, αντικατοπτρίζει κατά το ίμιση αυτά τα γεγονότα. Αναφέρονται ο Μλάντης, ο Κάρατζης, αλλά δεν βλέπω το όνομα μουσουλμάνων που κι αυτοί κάνανε εγκλήματα στη Σρεμπενίτσα σε αυτή την φοβερή διένεξη. Δεν βλέπουμε το όνομα του επικεφαλής μιας ε, ομάδας ε, στρατιωτικής των μουσουλμάνων που τα Χριστούγεννα το 1993 σε ένα χωριό χριστιανών έκανε εγκλήματα και δεκάδες χωριά καταστραφήκανε από τους μουσουλμάνους. Δεν το βλέπουμε ούτε αυτό στο κείμενο. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι και να επιβάλλουμε ε, διπλά με, ε, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ανάλογα με την περίπτωση υπάρχουν οι χριστιανοί που κάνανε εγκλήματα εις βάρος του αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το αντίθετο. Δεν έχουν επαληθευθεί ορισμένοι, ορισμένα εγκλήματα. Ε, έγινε στη Σερπενίτσα, έχουν εντοπιστεί μαζική τάφη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την άλλη πέρα που έχει διαπράξει εγκλήματα. Δηλαδή οι χριστιανοί τι ήταν, ζώα ήταν, πρέπει και αυτοί να αναφερθούν. Τι μπορεί να πει κανεί για δύο λεπτά όταν θέλουμε να περιγράψουμε αυτό που έγινε στη Σρεμπενίτσα και να μάθουμε πώ ακριβώ μπορούμε να θυμόμαστε για να μην ξαναπανληφθεί κάτι τέτοιο. Πολλά έχουν υποθεί για αυτό το γεγονό. Τι να πω εγώ που εγώ είμαι εδώ βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά γεννήθηκα στη Βοσνία τώρα εδώ ε, προσωπώ τη Σουηδία εγώ ε, κύριε Σιγιάνοφ μπορώ να σας πω αληθινές ιστορίες από εκείνη την περίοδο Αν κάποιο στην Ευρώπη είχε δει τι είχε γίνει, πραγματικά ο κόσμος θα είχε δράσει. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ τα γεγονότα. Θυμάμαι πεινασμένα παιδιά να φωνάζουν αίμα ε, εδώ και εκεί. Ένα κορίτσι να φωνάζει διότι έχει χάσει τους γονείς της. Έχω δει στρατιώτες να μεταφέρουν νεκρά πτώματα. Θυμάμαι το πρόσωπο του μπαμπά μου και θυμάμαι που ο ξάδερφός μου και άλλοι συγγενείς ήταν σε στρατόπεδο κεντρώσεις Και θυμάμαι κι άλλες ελλείψεις, αλλά θυμάμαι ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να ξεχάσω εκείνο το συνέστημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι οι τραγωδίες που έχει ζήσει κανείς γίνανε έτσι ανοιχτά και δεν μπόρεσε κανείς να εμποδίσει αυτές τις τραγωδίες. Κύριε Σογιάνοφ, ε, ε, θέλω να σας αναφέρω αυτά τα αισθήματα ενός θύματο στη Βοσνία που, που είναι ένα από τα θύματα σε όλα τα άλλα που έχουμε στα Βαλκάνια. και είναι γεγονός ότι οι Βόσνοι δεν θα ξανακερδίσουν ποτέ αυτούς τους αγαπημένους που χάσανε αλλά θα δώσει αυτό μια ευκαιρία σε εμά ε, να γίνει κατανοητό ότι η Ευρώπη έχει δει την τραγωδία μας και θα κάνει τα πάντα να μην ξαναπανεληφθεί αυτό. Εγώ δουλεύω ούτω ώστε η Στρεμπενίτσα μαζί με τη Βοσνία και οι άλλες βαλκανικές χώρες να γίνουν μέλη στην ευρωπαϊκή οικογένεια και θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα, να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα του η Ευρώπη να μην να δυνατή να αντιμετωπίσει τέτοιε καταστάσει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Νταϊάννα Γόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τα σχόλιά σα και για την ενίσχυσή σα προ την πρωτοβουλία αυτή. Τον προηγούμενο Ιούλιο είχα το πλεονέκτημα την υποχρέωση να παρευρεθώ στην ε, τελετή μνήμης της Ρεμπρένιτσα. Με σημάδεψε, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσω. Χιλιάδες ε, άνθρωποι είχαν μαζευτεί στον καύσωνα του ηλίου, αξιοπρεπείς, λυπημένοι, σε μια επέτειο τέτοια μνήμης και λύπης. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε, γιατί όλοι μας ως Ευρωπαίοι έχουμε μια αίσθηση τεζαβού για την καταστροφή αυτή. Μία αίσθηση συνενοχής. Όλοι είδαμε στις ίδιες μας τηλεοράσεις, στις κοινέ, πριν από τις φαγές, πριν από την πτήση στο τόρσο. Είχαμε αυτή την αίσθηση έλλειψης ελπίδας, έλλειψης ε, δυνατότητας αντίδρασης. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ξανά, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα θυμόμαστε, θα διδαχθούμε θα βοηθήσουμε τον κόσμο να προχωρήσει προς τα εμπρός. Και αυτό ακριβώς πρέπει να σημαίνει αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα επαιτίου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά που έζησα, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μητέρες, τις κόρες, τις γυναίκες, τις οικογένειες που γνώρισα εκείνη την περίοδο. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε κάτι που θα διαρκέσει για το μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ. να δώσω το λόγο στους ομιλητές στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ τώρα. Καταρχάς, η κυρία Πεζίσκα. Η 11η Ιουλίου ως μέρα μνήμης για τα θύματα της ε, Στεμπρένιτσα δεν θα πρέπει να μας κάνει να θυμόμαστε την ε, αναποτελεσματικότητα που είχε η διεθνή κοινότητα στο να προστατεύσει τα θύματα. Μετά από την πτώση της Σρεμπρένιτσα πάνω από 8.000 άνδρες και αγόρια σφαγιάστηκαν, 25.000 άτομα εκτοπίστηκαν και πολλές γυναίκες διάστηκαν. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε ποτέ αυτές τις πράξεις βίας. Ελπίζω όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν με αυτήν την ημερομηνία. Θα πρέπει να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα στεναρό προκειμένου να μην υπάρξει μια δεύτερη στρεμπένιζα. Και επίσης χρειάζεται να φροντίσουμε όσοι διαφεύγουν της σύλληψης να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Θα πρέπει να δούμε όσον αφορά τις σταθεροποίηση στα Βαλκάνια και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσει κανείς την ιστορία του. Το να θυμηθούμε την 11η Ιουλίου είναι μια συμβολική πράξη που εντάσσεται σε αυτό το πνεύμα. Εν μια απόδοση φόρου τιμής σε όλα τα θύματα και στις οικογένειές τους. Και μετά μια έκκληση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να δράσουν ούτως ώστε να απαυθούν τέτοια εγκλήματα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική η οποία να τις επιτρέπει να επέμβει εν ονόματι των ανθρωπιστικών αξιών. Και οι δυτικές βαλκανικές χώρες θα πρέπει να κάνουν τα πάντα ούτω ώστε να ενταχθούν στην δική μας οικογένεια. Αυτό σημαίνει όμως μια συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να στείλει. Ένα μήνυμα για το μέλλον. Και να διατηρήσουμε τις μνήμες μας ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκατσίν. Εγώ ήρθα σε επαφή με οικογένειες των θυμάτων και θα μου ζήτησαν να σας μεταφέρω τα ευχαριστήριά τους για την σημερινή συζήτηση. Και θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Αυτό το ψήφισμα δεν αφορά στο παρελθόν, μόνο ότι μιλάει για νεκρούς αφορά στους ζωντανούς και σε ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς. Ευχαριστώ. Boiul care a însoțit destrămarea fostei Iugoslavii reprezintă o pagină neagră în istoria Europei Uh, Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα παρατηρεί ο Πρόεδρος. Ναι, συνεχίστε να ελέγξουμε. Πρόκειται για ένα τραγικό ιστορικό γεγονός από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ότι χρειάζεται να είμαστε αποτελεσματικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική άμυνας ασφάλειας και στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα ό,τι φορά την πολιτική γειτονία για να καταπολεμήσουμε θέματα όπως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιφερειακές συγκρούσεις και παρά, παράλληλα παρόμοια φαινόμενα για η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια προληπτική πολιτική ώστε να μην επιτρέψουμε στο μέλλον παρόμοιες πράξεις. Ευχαριστώ. Και τώρα ας ακούσουμε το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε την σημαντική συζήτηση για τη Στρεμπρέντσα. Θα θέλω να σας διασφαλίσω ότι το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο πως οι δράστες ε, αυτών των ε, εγκλημάτων στην Στρεμπρέντσα, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, αλλά και οπουδήποτε αλλού στα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η αποστολή STP στην Βοσνία Ριζεγοβίνη συνεχίζει να ε, παρέχει βοήθεια στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο. Η Σεμπένιτσα ήταν και θα παραμείνει ένα πολύ σημαντικό παράγοντας ε, στην ζωή στην Βοσνία Ζεγοβίνη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη διεθνή κοινωνία. Θα πρέπει να κάνω έκκληση προς τους ηγέτες της Ζεγοβίνης να αποφύγουν το να αναφέρονται για πολλούς λόγους σε αυτήν την θλιβερή, σε αυτήν την οδυνερή ιστορική στιγμή. Θα πρέπει να φροντίσουν για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας της. Χρειάζεται λοιπόν να καλυφθούν προσπάθειες όχι μόνο στη Σρεβενίτσα αλλά και στη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο σύνολό της. Ε, Σρεβενίτσα συνέβη διότι δεν υπήρχε αρκετό ευρωπαϊκό πνεύμα και θα πρέπει τώρα να βοηθήσουμε την χώρα αυτή να ορθοποδήσει και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο βήμα ήταν η συμφωνία που υπογράφηκε με την χώρα για μια μακρά διαδικασία προσχώρησης, αλλά χρειάζονται περισσότερο, περισσότερο κουράγιο, περισσότερη εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να προωθήσουμε την συμφιλίωση όλοι έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και κυρία Ιμπρισάτσι. Ήμουνα μία από τα από τα άτομα εκείνα τα οποία έβλεπε τηλεόραση όταν συνέβησαν τα πράγματα, τα, οι φρικαλαιότητες αυτής. Και όλοι πιστεύαμε ότι ήταν ασφαλή το καταφύγιο, ασφαλές το καταφύγιο. Νομίζω ότι πραγματικά σοκαριστήκαμε όταν καταλάβαμε ποια ήταν η πραγματικότητα και όντως πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάθαμε από σκληρά παθήματα το τι θα πρέπει να κάνουμε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο και από εκεί συνεχίσαμε γιατί είδαμε ότι όταν δεν είμαστε ενωμένοι όντω συμβαίνουν τέτοιες φρικαλαιότητες. Και συνέβη αυτή η φρικαλαιότητα. Δεν μπορώ παρά να αποτίσω φόρο και σε εσάς που βρεθήκατε εδώ πέρα σήμερα μαζί μας που τόσο ανοιχτά μιλήσατε για τη συμφιλίωση. Ζείτε με τη μνήμη αυτή, θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι εκ παραλίλου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προπτική της Βοσνίας Αρζεγοβίνης να ενταχθεί στην Ένωση, ίσως αυτό να, μπορεί, να, είναι, να μπορέσει να αποτελέσει κάτι το οποίο θα συμφιλιώσει τη μνήμη με τις φρικτές αυτές φρικαλαιότητες. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος που έχουν εκτατεθεί από τις πολιτικές ομάδες. Ψηφοφορία των ε, ψηφισμάτων θα γίνει αύριο. Ήταν μακρά η συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους. Πέρα τη συζήτηση. Καλό βράδυ.